είναι δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικές ασφαλείας θέμα. Τουρκικές ενέργειες που προξενούν εντάσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Επίτροπο κύριο Χάν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Παρακολούθησα ε, εκ του και τα πρόσφατα γεγονότα στην ΑΟΣ της ε, Κυπριακής Δημοκρατίας και γενικότερα τις συνέπειες για την περιοχή. Γνωρίζουμε απολύτως τις ανησυχίες σας και τις επιστολές και τις ερωτήσεις που κάνατε πολλοί βουλευτές. Το πρώτο που θέλω να τονίσω σήμερα και να υπογραμμίσω είναι ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ' αυτού είναι πεντακάθαρη. Ε, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου έχει λεχθεί αυτό στην τελευταία έκθεση προόδου διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το επανέλαβε τον Οκτώβριο παρόλα αυτά έχει σημασία να επαναλάβουμε τη θέση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στεναρά υπέρ των κυριχειριακών δικαιωμάτων των κρατών μελών για διμερείς συμβάσεις και για εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων σύμφωνα με το κοινοτικό και εκτιμένο και το διεθνές δίκαιο συμπεριλαμβανομένο ε, σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρχουν απειλές, τριβές, προκλητικές ενέργειες που να βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ε, ειρηνική επίλυση διαφορών. Τώρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Περιμένουμε από την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΣ της, να δείξει συγκράτηση και να αποφύγει οποιασδήποτε δηλώσεις ή ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν και νέες τριβές. Είναι πολύ σημαντικό να μειωθεί η ένταση, να αποκλιμακωθεί προς όφελος όλων των μερών. Ταυτόχρονα ελπίζουμε η διερεύνηση και ενδεχόμενη εξόριξη και εξαγωγή φυσικών πόρων από την Κύπρο να μπορέσει να συνεχίσει και να είναι προς αμοιβέλο ε, όφελος όλων των Κυπρίων αυτό που δείχνει η σημερινή μας συζήτηση πάνω απ' όλα είναι η ανάγκη για ταχεία συνολική διευθέτηση του Κυπριακού μεταξύ των δύο κοινοτήτων, ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας. Δεν ήταν ποτέ τόσο επιτακτική αυτή η ανάγκη. Επ' θα ήθελα να ενθαρρύνω ε, έντονα και θερμά όλους τους ενεχομένους να συνεισφέρουν στο θετικό κλίμα και να οδηγηθούμε στην επίλυση του Κυπριακού προς όφελο όλων συνεχίζεται επί πολύ μακρόν ο διχασμός. Η επίλυση θα ανοίξει το έδαφος για τους φυσικούς πόρους ε, και θα έχει οικονομικά ε, ωφέλη ε, για όλους τους Κυπρίους. Οι επικεφαλείς των δύο κυπριακών κοινοτήτων έχουν επιδείξει και όραμα και θάρρος στις 11 Φεβρουαρίου με την κοινή δήλωση να ξαναρχίσουν τις ε, συζητήσεις. Το Σεπτέμβριο δεσμεύτηκαν να επιταχύνουν τις συνομιλίες. Τώρα καλώ και τις δύο κοινότητες και τους ηγέτες να βρουν έναν τρόπο να επιστρέψουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και να επαναλάβουν ουσιαστικές ε, διαρθρωμένες ε, διαπραγματεύσεις το συντομότερο, ανοίγοντας το δρόμο για μια δίκαιη, βιώσιμη και συνολική επίλυση του Κυπριακού προς όφελος των πάντων. Αυτό καλεί και ο ΙΕ. Έχουμε τον κύριο Μπαρτ Άιτερ που είναι ο εκπρόσωπος ε, του ΟΗΕ για την Κύπρο, ειδικό σύμβουλος και θέλει να βοηθήσει και τα δύο μέρη να γεφυρώσουν τις διαφορές, να επανέλθουν στις συνομιλίες και να κάνουν πραγματική πρόοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρά και στεναρά υποστηρίζει αυτές τις δραστηριότητες. Θα ήθελα να πω δύο λόγια γενικότερα για την Τουρκία. Ως μια χώρα ε, που έχει σταθερή ευρωπαϊκή προοπτική και δεδηλωμένη θα πρέπει να σέβεται τις υψηλότερες δημοκρατικές προδιαγραφές και πρακτικές ανεπιφύλακτα. Ε, θα ε, τη ζητήσουμε ένα λογοδοτήση γι' αυτό και εμείς θέλουμε να έχουμε ε, ενισχυμένες ε, και πιο βαθιές σχέσεις με την Τουρκία και είναι και προσωπική μου πρόθεση. Αυτό σημαίνει όμως και ευρύτερη σχέση, ε, πολιτικό διάλογο, καλύτερη συνεργασία Έχουμε πολλές κοινέ προκλήσεις στην περιοχή. Μια πιο ε, παραγωγική και πιο στενή και οικονομική σχέση υπέρ των πολιτών μας μέσω της εμβάθυνσης της ε, Τελωνιακής Ένωσης. Και περαιτέρω πρόοδος χρειάζεται για ε, θέματα μετανάστευσης και απελευθέρωσης θεωρήσεων διαβετηρίων. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να ενισχύσω και να συσφίξω τους δεσμούς με την Τουρκία προς όφελος όλων και αμοιβαία ευεργετήματα. Ε, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα και πάλι να σας διαβεβαιώσω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ ψηλά στις δικές μου προτεραιότητες. Παρακολουθώ από στενά τις εξελίξεις, κατανοώ τις ανησυχίες σας. Σήμερα στην Άγκυρα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και οι ψηλοί παράγοντες έχουν συνομιλίες. Ε, το θέμα αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη, καθότι υπάρχει αίσθηση του επίγοντος να προχωρήσει το Κυπριακό και να επιληθεί. Και θα παρακαλούσω και την τουρκική κυβέρνηση να δει πώς μπορεί να βοηθήσει για να βελτιωθεί η κατάσταση και οι σχέσεις. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ε, περιμένω να ακούσω τις απόψεις για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπο, λέει Πρόεδρος. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, με πρώτο τον κύριο Μπρόκ, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Παρακαλώ κύριε Μπρόκ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κύριε Πίτροπε, σωστά τα είπατε. υπάρχει τεράστια δυνατότητα για όλες τις χώρες στην περιοχή. Δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο ανόητοι, γιατί στην ανθρωπότητα συχνά το κάνουμε. Τσακωνόμαστε για διάφορα θέματα και τελικά δεν κερδίζει κανένας και ε, έχουμε πολέμους. Το καλύτερο είναι να συζητούμε μεταξύ μας, να διευθετούμε τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχει το διεθνές δίκαιο που πρέπει να ισχύει. Και κατανοώ τους ε, πρίους βουλευτές ε, που λέγουν ότι όταν στα χωρικά τους ύδατα ε, κάνουν ε, ε, διερεύνηση και προχωρούν σε γεωτρήσεις. Έρχεται η Τουρκία και τους παρενοχλεί και είτε είναι μέλος της Ούγκλος είτε δεν είναι. Αυτό δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει και ε, είπανε και η επίσημη η κυπριακή κυβέρνηση ότι θα είναι προς όφελος και των δύο πλευρών οι πόροι. Δεν είναι μόνο για το ελληνικό τμήμα, είναι για όλους τους κατοίκους της Κύπρου. Γι' αυτό και ε, θα πρέπει να το καταλάβει και η τουρκική κυβέρνηση. Ε, είναι θέμα διεθνούς δικαίου που θα πρέπει να εφαρμόζεται και να υλοποιείται. Αλλά στα πλαίσια μεγάλης συνεργασίας και ειλικρίνειας με συζήτηση και να αποσκοπούμε όλοι σε μια κοινή λύση για να λυθεί πρώτα αυτό το ζήτημα το κυπριακό που έχει να κάνει με τη διχοτόμηση της νήσου και να επανενωθεί και να είναι ενωμένη αλλά γενικότερα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα και είναι και ένα ζήτημα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θέλουμε να διαφοροποιήσουμε και ε, τις ενεργειακές πηγές και θα ήταν ανόητο να μην λυθεί αυτό το θέμα. Έχει συμφέρον και η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ε, είμαστε στο πλευρό και των Κυπρίων συναδέλφων που έχουν δίκιο, αλλά να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση και στις συνομιλίες με την Τουρκία και να προχωρήσουμε προς μια ειρηνευτική προσπάθεια και ειρηνική επίλυση του θέματος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπρόκ. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο για την πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε επαναλαμβάνοντας ένα χωρίο του ψηφίσματο το οποίο αύριο πρόκειται να εγκρίνουμε. Ανησυχούμε πάρα πολύ όσον αφορά την παρουσία της ε, Τουρκία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ενό μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κύπρου. Θα πρέπει αυτέ οι ενέργειε να σταματήσουν πάρα Ζητούμε από την Τουρκία να σεβαστεί τι υποχρεώσει τι οποίε ανέλαβε ε, εναντί του διεθνούς δικαίου, αλλά επίση όσον αφορά και το καθεστώ που την διέπει ω υποψηφίου ε, μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και σταθμίσουμε τι συνέργειε στα χωρικά δέντρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά θέλω να σα πω από πλευρά τη πολιτική μα ομάδα, γιατί εμεί χωρί καμία επιφύλαξη θέλουμε ε, την ε, προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχει διάλογος με τους Τούρκους ομιλητές μας, θα συνεχιστεί και πρόκειται να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές. Πρόκειται για στρατηγική σημασία χώρα για εμά και για αυτό τον λόγο, άπαξ και η Τουρκία ε, θέλει να έχει ε, σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και εγγυήσει για ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Τώρα, ε, κατά θέλω να σας πω ότι η πολιτική μας ομάδα υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις για την επανένωση των δύο μερών της Κύπρου των δύο τμήματων τέλο πάντων και όσον αφορά την εκμετάλλευση των ε, υδρογοναδράκων, αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και για τις δύο κοινότητες για όλη την Κύπρο αλλά και τις υπόλοιπες χώρες που εμπλέκονται ευχαριστούμε πολύ λέει η πρόεδρος και τώρα για τους μεταρρυθμιστές ε, συντηρητικούς και το λόγο κύριο Στάνοκ ο λόγο ότι πήγε εκεί πέρα η Τουρκία και εισέβαλε σε αυτή την αόζη είναι αυτό κατάφορη παραδείγμα του διεθνού δικαίου. Σύμφωνα με το δίκαιο τη θάλασσα, πρόκειται για μια ε, πράξη απαράδεκτη και επομένω την διαδικασία τη επανένωση έτσι την πυροδοτούν οι Τούρκοι και την δυναμητίζουν. Οπότε το θέμα είναι τι θα έκανε η κυβέρνηση. Φυσικά και θα σταματούσε τι συνομιλίε. Επίση, βέβαια, δεν πρέπει να συμφωνήσουμε ε, με αυτό το οποίο είπε η γύρω ότι δεν θα πρέπει, αν δεν υπάρχει κάποια οριστική ρύθμιση, να αποφασιστεί ότι θα γίνει με τους γιατί έχουμε επανειλημμένες ε, διαβεβαιώσει ότι πρόκειται όλοι να ωφεληθούν από το φυσικό αέριο. Αυτέ είναι διαβεβαιώσει και αυτέ οι διαβεβαιώσει όμω θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές ως καλόπιστε και από του Τούρκου. Το, τα έσοδα από τα κοιτάσματα αυτά πρόκειται να ωφελήσουν και τι δύο πλευρέ και πρόκειται να είναι ένα κίνητρο ούτω ώστε να προωθηθούν, να προχωρήσουν οι συνομιλίε. Θα πρέπει επίση να αποδοθεί η, η αμόχθος και αυτό θα ήταν μια κίνηση καλή πίεσης από πλευράς ε, Τούρκων. Ε, επίσης το ούγκλος θα πρέπει να εγκριθεί, ε, να αγκαλιαστεί από το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές και θα πρέπει και η Τουρκία να ξαναθυμηθεί τις δεσμεύσει της όσον αφορά τη Συμφωνία της Άγκυρας αλλά επίση και τις υποχρεώσεις της ως υποψηφία χώρα και έτσι ε, να ε, αναγνωριστεί και από τις 28 χώρες αλλά και από την η Τουρκία και τις 28 χώρες και την ε, Κυπριακή Δημοκρατία. Το λόγο τώρα έχει εξ όνομα της ομάδας το κύριος Βαν Μπάλεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομάδα Άλντε δεν θέλει να διωγγώσει το πρόβλημα, αλλά να το συρρυκνώσει. Πώς θα γίνει αυτό? Μόνο παραπέμποντας στο διεθνές δίκαιο. Και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, η αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν έχει καμιά δουλειά εκεί μέσα η Τουρκία. Μπορεί μόνο να εξερευνεί ε, κανείς ή να εκμεταλλεύεται μόνο με την άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας εκεί. Ξέρω, καταλαβαίνω αυτά που λέτε ότι οι δύο κοινότητες δεν θα πρέπει απλώς να συμφωνήσουν αλλά και να υποφελούνται από τους φυσικούς πόρους. Για να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει, Άρα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κρατηθεί στο και να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί η Τουρκία να συνεχίσει τις δραστηριότητε τη στην ΑΟΣ της Κύπρου. Τέλεια και Παύλα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει εξ ονόματος της ομάδας της η κυρία Γκάμπη Τσίμερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας να καταδικάσω σποδρότατα τις σεισμικές έρευνες που κάνει η Τουρκία στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και καλό και την Τουρκία αμέσως να πάψει αυτές τις δραστηριότητες. Και ξέρουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το βόρειο-δυτικό τμήμα της ε, Κύπρου. Τώρα όμως είναι στην νότια ακτή. Τι δουλειά έχει εκεί πέρα η Τουρκία. Και μέχρι τώρα ε, δεν ε, έχει προβάλει καμία αξίωση για αυτά τα ύδατα και είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφανθεί και σωστά αναμένουν και οι Κύπροι φίλοι και συνάδελφοί μας να ε, εκφράζονται τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και οι διεθνείς οργανισμοί και να μην σιωπούν και να το αποδέχονται σιωπηρά. Πόσο μάλλον που διαπραγματεύσεις για την ευρύτερη λύση του Κυπριακού έχουν ανασταλεί. Η Τουρκία προκάλεσε την κρίση, η Τουρκία έχει και την ευθύνη για την αποκλιμάκωση ε, και την ε, καταστολή και τον κατευνασμό για να επανέλθουν οι συνομιλίες. Και θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό υπήρξε μία πρόταση του Δημήτρη Χριστόφια με τον κύριο Ταλάτ να συμφωνήσουν για την ε, θαλάσσια ζώνη. Περί τίνος πρόκειται. Ε, αυτές οι ζώνες ε, είναι ομοσπονδιακή αρμοδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτό θα ίσχυε και για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Δυστυχώς αυτές οι διαπραγματεύσεις βάγισαν ε, από τον κύριο Έρογλου ε, τον αντικαταστάτη και διάδοχο του κυρίου Ταλάτ. Λοιπόν, το Κοινοβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε να επιμείνει να βρεθεί λύση του Κυπριακού προβλήματος, γι' αυτό ε, ζητούμε και να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο και υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες που ε, οδηγούν σε μια λύση διζωνική με ισότητα για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Σκρόλετς, εξ ονόματος των Πρασίνων. Έχετε ένα μισό λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε Χάν, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να πω ότι ανησυχώ με όσα έχουν ε, προκύψει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Τα γεγονότα αυτά ε, έχουν πάψει κάθε ε, ειρηνευτικές, τις διαπραγματεύσεις της ειρηνευτικές. το δίκαιο της θάλασσας παραβιάστηκε. Η Κύπρος είναι κατός μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό λοιπόν να φροντίσουμε για να αποκατασταθεί ένα θετικό κλίμα και για τις δύο πλευρές. Η αναζήτηση υδρογονανθράκων και καυσίμων στην ε, αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου είναι κάτι που αφορά ε, προφανώς και την Ελλάδα και την Κύπρο και βεβαίως η ανακάλυψη τέτοιων κοιτασμάτων θα είναι πολύ σημαντική για, για ολόκληρη την ίσο. Πρέπει λοιπόν η συζήτηση για τις συμφωνίες αυτές να επιτρέψει να δημιουργηθεί ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους κατοίκους της νήσου. Παρά τις πολιτιστικές και θρησκευτικέ διαφορές που ανέκαθεν υπήρχαν, αλλά ουσιαστικά αποτελούν το πολιτιστικό πλούτο της Κύπρου και ολόκληρου του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η συνέχιση λοιπόν των διαπραγματεύσεων και το να βρεθεί μία λύση για, τις, για όλες τις αντιφερόμενες πλευρές είναι στρατηγική σημασία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Τουρκία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αφρόντε. Έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτή τη στιγμή, στα ύδατα τη Κύπρου υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ τη Τουρκία και τη Κύπρου για την ενεργειακή ασφάλεια. Πόσε φορέ δεν είπαμε ότι στην Ευρώπη θέλουμε μια ένωση λαών που να ενωθούν. Θα πρέπει να δούμε ότι η Ευρώπη δεν είναι απλώ μια ένωση προσώπων και να μην είναι αδύναμοι οι κανόνε με του οποίου έχουμε οπλιστεί. Θα πρέπει να μην επιτρέψουμε τη σύγκρουση αυτή ε, να συνεχιστεί. Η Κύπρο θα πρέπει να προστατευτεί, αλλά αυτό δεν έγινε. Χθε προέκυψε μια μελέτη που δηλαίει ότι 30% των Κυπρίων δεν αισθάνονται ότι είναι μέρος ε, της, ε, μάλλον θα πρέπει να είναι με φυσικό τον τρόπο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι αισθάνονται. Και μιλάμε και για ε, ένα κράτος που έχει κυρώσει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αλλά και η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν αναγνωρίζει ένα άλλο κράτος μέλος αμφισβητεί τα χωρικά του ύδατα. Μιλάμε για ένα ε, νησί το οποίο είναι χωρισμένο στα δύο με την κατοχή από, από στρατεύματα και θα πρέπει με πυγμή να επιβεβαιώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει με μια ενιαία φωνή εξ όλων των κρατών μελών της, πατάσσοντας αυτήν την συμπεριφορά. Ε, ε, Ο κύριος τώρα. Έχετε ένα λεπτό. Ο κύριος... Αποτελεί έσχο το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση τη Κύπρου εθελοτυφλεί. Δεν υπάρχουν δύο κοινότητε. Υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Εδώ και 40 χρόνια χαϊδεύουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί την Τουρκία η οποία κατέχει αυτή τη στιγμή το 37% του ευρωπαϊκού Εδάφου, δηλαδή τη κυπριακή Δημοκρατία. Κατέχεται όμω παράνομα από την Τουρκία που έχει και το θράσο να χτυπά την πόρτα τη Ευρώπη μιας χώρας που δεν συμμορφώνεται με τα ψηφίσματα του συμβουλίου ασφαλείας του οηε που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο με επίκηση των κατεχομένων που επικαλείται το δίκαιο της θάλασσας το οποίο δεν έχει υπογράψει καν που ενάντια σε κάθε λογική ηθική και νομική διάσταση θεωρεί ότι μπορεί να καταπατά κυριαρχικά δικαιώματα άλλου κράτους. και εμείς συζητάμε για λογικές διευθετήσεις ενώ προχωρήσαμε κόντρα σε κάθε λογική σε κυρώσει κατά της ρωσίας. τι συζητάμε λοιπόν αντί να πράττουμε; οι τουρκικές ενέργειες στην αός της κύπρου συνιστούν άμεση επιθετική ενέργεια κατά της ευρωπαϊκής ενώσεως. καμία συζήτηση και ενέργεια μέχρι η τουρκία να αποσύρει το ερευνητικό σκάφος και τα πολεμικά πλοία από την περιοχή να προχωρήσει σε κατάργηση του ψευδοκράτους και να αναγνωρίσει επίσημα την κυπριακή δημοκρατία. ήδη η τουρκία έχει αποκαλύψει το πραγματικό της αυτό σε ό,τι αφορά τους τζιχαντιστές του ισλαμικού χαλιφάτου. μια υπερφύαλη επεκτατική και επιθετική χώρα μπαμπούλας με σύνδρομα οθωμανισμού του παρελθόντος. επιτέλους είναι καιρός να πάψουμε να την ανεχόμαστε. επιτέλους ας Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Θεοχάρου. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε θίξει πολύ σημαντικέ πτυχέ του προβλήματο τη Κύπρου και σα ευχαριστώ θερμά. Κύριε Επίτροπε, σας επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι το πρόβλημα δεν είναι μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Το πρόβλημα είναι η Τουρκία, η οποία παράνομα κατέχει στρατιωτικά με τη δύναμη των όπλων της εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτή τη στιγμή επιχειρεί να καταλάβει και τις θάλασσες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ενέργειες της Τουρκίας έχουν κριθεί ως παράνομες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, από ευρωπαϊκά δικαστήρια. Μας είπατε πριν από λίγο από την Επιτροπή, από το Συμβούλιο, η Τουρκία δεν καταλαβαίνει από εκκλήσεις κύριε Επίτροπε. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε εκκλήσεις τη στιγμή που ο άλλο στέλνει τα θωρακτά και τα υποβρύχια του μέσα στην θάλασσα της Κύπρου εκείνο που ζητάμε είναι να καταδικαστεί η τουρκία και να ληφθούν πρακτικά μέτρα εναντίον της οικονομικές και πολιτικές κυρώσεις και να ανασταλούν οι ενταξιακές συνομιλίες σύμφωνα με την δήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου με την οποία είναι δεσμευμένη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Τουρκία ορθώνει ένα τείχος χειρότερο από το τείχος του Βερολίνου και χωρίζει τον λαό της Κύπρου στα δυο και χωρίζει τα εδάφη της Κύπρου στα δυο. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε αυτή την πραγματικότητα και να βοηθήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία να σταθούμε αλληλέγγυοι στην Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη δύναμη των όπλων. Τα όπλα δεν δημιουργούν δίκαιο κύριε Επίτροπε. Τα όπλα μόνο παρανομία επιβάλλουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα κύριος Χάουιτ για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω απολύτω με τους Κυπριούς συναδέλφους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών που λένε ότι απειλείται η εθνική τους κυριαρχία και ότι θα πρέπει να ισχύσουν οι κανόνε του διεθνού δικαίου. Συνυπογράφω το ψήφισμα αυτό και πρέπει να πω στου Τούρκου φίλου ότι εμεί εδώ μαζί με τον ε, Επίτροπο Χαν θα πρέπει να δείξουμε, θα δείξουμε πυγμή και θα πρέπει να πάψει οποιαδήποτε περαιτέρω δράση που μπορεί να προκαλέσει τριγμού. Θα πρέπει όμω ο Επίτροπο ε, στην ομιλία του ε, να δει πώ εννοεί την ευρωπαϊκή προοπτική τη Τουρκία όπω την ανέφερε και την ειδική σχέση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Το Κοινοβούλιο δεν περιέλαβε στο κοινό αυτό ψήφισμα και δεν ε, έχει αναφερθεί αρκετά στην ε, στο σχετικό εδάφιο την δέσμευση να συνεχιστούν οι συνομιλίες ε, για την ενοποίηση και την εξέβρεση λύσης, την ερνευτική διαδικασία για το πρόβλημα του Κυπριακού. Θα πρέπει να πω ότι πάντοτε επιδεικνύω αλληλεγγύη προς τους Κυπρίους συναδέλφους, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να προωθηθεί η συμφιλίωση, να υπάρξει οικοδόμηση εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών και αναγνωρίζοντα την ανάγκη εξέβρεση διπλωματική λύση για να λυθεί η τρέχουσα κρίση και να πάψει ο διαμελισμό τη νήσου. Οι εμπορικέ ε, δραστηριότητε και η αναζήτηση υδρογοναθράκων είναι κάτι που θα πρέπει να ωφελήσει και τι δύο κοινότητε τη Κύπρου. Θα ζητήσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν τη θέση αυτή και να στηρίξουν την δική μας τροπολογία. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να δείξει πειθαρχία το Κοινοβούλιο και να μην επιτρέψει να συνεχιστούν οι προκλήσεις, αλλά να επιδιώξουμε την αποκλιμάκωση προς συμφέρον όλων. Σας ευχαριστώ, συναδελφέ Χάουιτ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πανόρντον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι θέλουμε μία λύση για το Κυπριακό και οι δύο πλευρές ε, φέρουν κάποια ευθύνη αναμφίβολα για την τρέχουσα κατάσταση, αλλά με πάσα ειλικρίνεια δεν βοηθάει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο να ξαναξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για ένα μονομερές ψήφισμα που θέλει να δώσει όλο το φταίξιμο στην Τουρκία, στους Τουρκοκυπρίους ή ο Επίτροπος να μιλάει με τον τρόπο που μίλησε στην αρχή και Ελπίζω να με ακούει τουλάχιστον τώρα. Δεν νομίζω να με ακούει. Με ακούτε. Επίτροπε. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι φορά το πρόσφατο αντιέξοδο θα πρέπει να κοιτάξουμε στα αίτια, να τα ζητήσουμε στο 2004. Το Μάιο η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησε να μπλοκάρει οποιαδήποτε πρόοδο, ιδιαίτερος σε ό,τι αφορά το εγχείρημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον προηγούμενο μήνα να, να τερματιστεί η απομόνωση της Βόρεια Κύπρου. Αν είχαν τηρηθεί αυτές οι δεσμεύσεις, καμία από τις δυσκολίες που συζητούνται σήμερα δεν θα είχε προκύψει. Κύριε Φανόρντεν, μία ενδιάμεση ερώτηση, μία ερώτηση από τον κύριο Χατζηγεωργίου. Δέχεστε. Ε, δεν θα πω ότι ο κύριος Βανόρτεν είναι προκλητικός, αλλά ε, θα κρίνω ότι είναι από άγνοια. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, έχετε διαβάσει την συμφωνία μεταξύ Χριστόφια Ταλάτ που λέει ότι αυτά τα αποθέματα ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία που θα είναι ομόσπονδη μετά τη λύση, αν το έχετε διαβάσει αυτό, και αν ξέρετε επίση τη συμφωνία πάλι Χριστόφια με τον Νερογλου, τον οποίο υπερασπίζεστε ασμένος, είναι ένας διχοτομιστής όμως, η οποία συμφωνία καθορίζει και τον τρόπο διαμοιρασμού, ποσοστιαία δηλαδή. Ε, εν πάση περιπτώσει, το να είναι κανεί ευρωβουλευτή πρέπει να διαβάζει πριν ομιλεί. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Φανόρντεν. Όπως ο συνάδελφος και φίλος Γεωργίου θα γνωρίζει πολύ καλά, χαίρομαι να εξετάσω σε βάθος και λεπτομέρεια αυτά τα ιδιαίτερα θέματα και θα έλεγα ότι κανένα από το πρόβλημα αυτό αυτή δεν ήταν η συζήτηση σήμερα το απόγευμα, σήμερα το βράδυ. Πρόκειται για μονομερή κριτική της Βόρεια Κύπρου και της τουρκικής θέσης. Αν θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος για να ενωθεί η νήσος, όπως όλοι είμαι σίγουρος ότι θέλουμε. Η μοναδική λύση, από ό,τι ξέρουμε, είναι μια λύση που θα σεβαστεί τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα και των δύο κοινοτήτων στην νήσο. Και αυτό επανέρχεται στο σημείο που ανέφερα, αυτό που συνέβη το 2004. Και πολύ απλά πρέπει να το ξεπεράσουμε και πρέπει να μιλήσουμε με πιο γενναιόδωρο και ε, τρόπο που να δείχνει συμπάθεια προς τους ε, Τουρκοκυπρίους. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Φανούρτεν. Έχω διάφορες ε, ενδιάμεσες ερωτήσεις. Πολύ λυπάμαι, αλλά σήμερα το απόγευμα είχαμε μία έκτακτη συζήτηση και αυτό λοιπόν έχουμε καθυστερέσει πολύ. Έχουμε αντιπρόεδρο που δεν μπορεί να φτάσει μετά τα μεσάνυχτα. Θα είμαι πολύ αυστηρός λοιπόν. Θα επιτρέψω άλλη μία ερώτηση, αν το είναι αποδέχεται ο κύριος Φανόρντεν, από την συνάδελφο Θεοχάρους και στη συνέχεια θα επιτρέπω μόνο μία ερώτηση. Η κυρία Θεοχάρους. Κύριε Φανόρντεν, συχνά κατηγορείτε τους Ελληνοκύπριους γιατί απέρριψαν το σχέδιο ΝΑΝ το 2004 και αυτό το κάνετε έμεσα σήμερα. Ξέρετε ότι οι Τυρκοκύπροι επίσης απέρριψαν το σχέδιο ΝΑΝ και όχι μόνο οι Ελληνοκύπριοι Οι επικιστές ήταν αυτοί που ψήφισαν υπέρ του σχεδίου Ανάν. Ο συνάδελφο Φανόρδεν, η απαντήση. Δεν ανέφερα το σχέδιο Ανάν. Μιλούσα για αυτό που συνέβη το 2004 και αναφέρθηκα πολύ συγκεκριμένα στην υπόσχεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2004 να τερματιστεί η απομόνωση της Βορειοκύπρου. Κύπρου. Ένα μήνα αργότερα όλα αυτά παραμερίστηκαν και έχουμε σημειώσει πολύ μικρή πρόοδο έκτοτε κάθε τρεις και λίγο μας δίνουν λίγη ελπίδα. Κάτι συμβαίνει που μας κάνει να πιστεύουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει πρόοδος και μετά ε, δεν γίνεται τίποτα. Θα πρέπει να το ξεπεράσουμε λοιπόν αυτό και να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε που θα κάνει σεβαστές τις ε, επιθυμίες όλων των πλευρών. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Φανόρντεν. Σας παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο ομιλία στο μέλλον για λόγους συναδελφικότητας. Ο συνάδελφος Κούζο Περμούη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι η δεύτερη φορά στην Ολομέλεια που χρειάζεται να αναφερθώ στις παραβιάσεις ε, του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία. Αυτή τη φορά όμως δεν μιλάμε για ε, πιθανή χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων ούτε πράξεις αποσταθεροποίησης ε, στη Μέση Ανατολή. Εδώ μιλάμε για απειλές της Τουρκίας σε μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στην Κύπρο. Οι τουρκικές ε, απειλές ε, από την Τουρκία που είναι χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ένωση, σας υπενθυμίζω, είναι απειλές προς όλους μας, προς όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετακινούνται στρατιωτικά, μάλλον ε, τουρκικά πλοία στα χωρικά ύδατα της Κύπρου. Έχουμε την οδηγία ΝΑΒΕ, την οποία έχουν παρανόμως εκδώσει οι ενόπλες τουρκικές δυνάμεις και παραβιάζει την νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν, είπατε εκπρόσωπος, ε, να είναι απερίφραστη στην καταδίκη της για τις καταδίκες του διεθνούς, της του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία και θα πρέπει να αναστείλει και τις ανταξιακές διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ στον αδελφό Κούζο και τώρα ένα λεπτό κύριος Καστάλτο. Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, δεν την καταλαβαίνω την Τουρκία, πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Μιλάμε για μια υπέροχη χώρα που εδώ και 30 χρόνια θέλει να γίνει μέρο τη Ευρώπη. Και σε αυτό το σώμα θα θέλαμε να μπορούμε να επενέσουμε την πρόοδό τη προ την προσχώρηση και το πόσο καλά χρησιμοποίησε τι ε, χρηματοδοτήσει που έλαβε. Κι όμω το αντίθετο συμβαίνει. Πρέπει να καταδικάσουμε το κλείδωμα και την πίεση που έχουν δεχτεί τα κοινωνικά δίκτυα. Επίση την οπορτονιστική αδιαφορία τη μπροστά στι φαγέ του Κομπάνε και τέλο την παράνομη εισβολή τη στην ε, οικονομική αποκλειστική ζώνη τη Κύπρου. Τι δρόμο είναι αυτό που έχει πάρει η Τουρκία. Εδώ δεν διακυβεύονται μόνο οι εξορίξει ανθράκων στη Μεσόγειο, ε, με τι οποίε εμεί από το Τσίνκου Εστέλε είμαστε ούτω ή άλλω αντίθετοι. Αλλά υπάρχει βαρύτατη ευθύνη τη καταστροφή των έφραυτων διαπραγματεύσεων μεταξύ τη Δημοκρατία τη Κύπρου και τη Βόρεια Κύπρου. Μια υποψήφια χώρα θα έπρεπε συνεπώ να μα βοηθήσει να ε, σβήσουμε μαζί την πυρκαγιά στη Μέση Ανατολή και να υπάρξει μια ίση κατανομή όλων των ευκαιριών για όλου του Κυπρίου. Να υπάρχουν ειρηνευτικέ και επικοδομητικέ διαπραγματεύσει. Όμω η, Ευρωπα... η Ένωση δεν γίνεται με τα ωραία λόγια, γίνεται μόνο με τι πράξει. Σα ευχαριστώ, συνάδελφε Καστάλδα. Και τώρα ο συνάδελφο Φεράν για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιουνκέρ που μας έκανε να καθυστερήσουμε δύο ώρες στη συζήτηση. Αυτός έφυγε και τρώει τώρα και εμείς ε, μένουμε εδώ. Έχουμε να συζητήσουμε όμως σοβαρά θέματα. Ποιο είναι το ε, ζήτημα απόψε, ε, ο κύριος Γιούγκερ ή η Τουρκία. Απευθυνόμενος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πράγμα έχω να πω μόνο. Απόψε μα στέλνετε να συζητήσουμε αυτό το θέμα χωρίς να έχετε κάνει εσείς ποτέ τίποτε για την Κύπρο. Χύνεται κροκοδίλια δάκρυα για μια ακόμη φορά χωρίς να υπάρχει καμία πρόοδος. Ε, επί της ουσίας, θέλω να πω ότι είμαστε υπερ ε, ισορροπημένων και δίκαιων διεθνών σχέσεων μεταξύ κυρίαρχων κρατών. Βεβαίως, ε, στόχος μας είναι η προάσπιση και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, που είναι εθνική αρμοδιότητα. Σήμερα όμως θα πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλα τα κράτη αυτές οι ζώνες και από την Τουρκία που, έχει υπογρά μάλλον που δεν έχει υπογράψει α, τη σύμβαση αυτή. Ιδίω σήμερα τίθεται, είναι στην επικαιρότητα η Κυπριακή Δημοκρατία και διακόπτεται ο μιλητής. Ο συνάδελφος Κεφαλογιάννης. Η τουρκική επιθετικότητα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου συνιστά κατάφορη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Η Τουρκία πρέπει να δεσμευτεί στις αρχές που διέπουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ όλων των κρατών του κόσμου. Η Τουρκία πρέπει να υπογράψει και να επικυρώσει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου, είναι η μόνη χώρα που εδώ και 20 χρόνια δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη UNCLOS που έχει ψηφιστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τέλος, η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στην υφαλοκρηπίδα όσο και στην αποκλειστική του οικονομική ζώνη. Η υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη των κρατών μελών είναι η υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Κεφαλογιάννη και τώρα η συνάδελφος πήρε για 1,5 λεπτό. Α, λεπτό κυρία Πύρη, συγχωρέστε με, ο συνάδελφος Ντάρτμορ θέλει να κάνει ερώτηση. Κυρία Κεφαλογιάννη, αποδέχεστε την ερώτηση. Αποδέχεστε την ερώτηση κύριε Κεφαλογιάννη. Πείτε. Sorry, uh, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Κεφαλογιάννη, είσαστε πάρα πολύ γλαφυρός σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις της Τουρκίας, σε ό,τι αφορά τη ε, Κύπρο και το δίκαιο της θάλασσα. Και θα γνωρίζετε κατά πάσα πιθανότητα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει πάνω από 900 εκατομμύρια κάθε χρόνο σε χρηματοδότηση προενταξιακή στην Τουρκία και ανάλογα κονδύλια έχουν προαξανακληθεί για τα επόμενα πέντε χρόνια. Είσαστε υπέρ των ποσών αυτών να συνεχιστούν. Και διακόπτει ο Σα Σα ευχαριστώ, συνάδελφε Ντάκμαθ. Ο συνάδελφο του Κεφαλογιάννη. Εγώ προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, θα ήμουν εναντίον να συνεχιστούν αυτά τα κονδύλια. Αλλά θα πρέπει να ξέρει ο κύριο συνάδελφο ότι αυτά δεν είναι θέματα τα οποία συζητούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι θέματα των ευρωπαϊκών συνθήκων τα οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Κεφαλογιάννη. Και τώρα το λόγο έχει η συνάδελφο Σπύρη. Πριν από 8 μήνε, το Σώμα καλωσόρισε τι θετικέ εξελίξει στην Κύπρο. Το κοινό ψήφισμα από του ηγέτε των ελληνικών και ε, κυπριακών κοινοτήτων τη της Κύπρου μιλούσαν για μια μελλοντική ενοποίηση της νήσου παρά τα ενεπίλητα προβλήματα που θα συζητούνταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να υπάρξει μια βιώσιμη και ειρηνική λύση. Τώρα όμως η θαλάσσια εισβολή της. Ε, Τουρκίας, την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας, έχει οδηγήσει στη διακοπή των αρνητικών συνομιλιών. Χάσαμε το ρυθμό που είχαμε πριν από 8 μήνες πλήρως. Αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο για τους κατοίκους της νήσου, αλλά θα επηρεάσει αρνητικά ολόκληρη την γεωγραφική αυτή περιοχή. Αυτό που χρειάζεται πάνω από όλα Ανατολική Μεσόγειος αυτή τη στιγμή είναι μια ακτίδα, ακτίνα ελπίδας και θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τι ευθύνε του. Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί τα δικαιώματα κυριαρχία τη Κύπρου και την αποκλειστική οικονομική τη ζώνη. Η νομιμότητα τη ζώνη αυτή δεν μπορεί να αμφισβητείται. Επίση, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η αιρεσιμότητα δεν μπορεί να ε, ε, εφαρμόζεται διαφορετικά στι δύο κοινότητε τη νήσου. Θα πρέπει όλοι να ωφεληθούν από τα κοιτάσματα αερίου. Θα πρέπει λοιπόν οι ηγέτε των δύο να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να βρουν μία μόνιμη λύση στο όλο πρόβλημα. Και το ίδιο και ο σύμβουλος, ε, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Άιντερ, το ίδιο τόνισε στις δηλώσεις του. Πριν από 8 μήνες οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων ε, δεσμεύτηκαν να αποφύγουν τον επονιδισμό και τις αλληλοκατηγορίες. Τώρα θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξει πάυση αυτής της προσπάθειας. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Πύρη και τώρα ένα λεπτό ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία έχει εισβάλει παράνομα στην Κύπρο και κατέχει παράνομα το 37% του κυπριακού εδάφους. Τώρα άρχισε να πραγματοποιεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και παράνομες σεισμολογικές έρευνες στην ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα της Κύπρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει αυστηρά μέτρα κατά της Τουρκίας, προκειμένου η Άγκυρα να σταματήσει την επιθετικότητά της απέναντι στην Κύπρο, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα το κοινοβούλιο μας πρέπει να διαμηνήσει στην τουρκία ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα της κύπρου να συνάπτει συμφωνίες για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στην ΑΟΣ δεύτερον να ζητήσει την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής. τρίτον να καλέσει την τουρκία να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να σταματήσει τις παράνομες δράσεις και απειλές κατά ιουδήποτε κράτους της ευρωπαϊκής ένωσης τέταρτο να πάψει η τουρκία να προβαίνει σε ενέργειες που αμφισβητούν το δικαίωμα της κύπρου να εκμεταλλεύεται τους υδρογονάνθρακες που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Μαριά και τώρα η κυρία Σακοράφα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθώντας την ερμαφρόδιτη πολιτική της διεθνούς κοινότητας στο Κυπριακό κατέληξε να διαπραγματεύεται την ένταξη της χώρας που με 45.000 στρατιώτες κατέχει 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ευρωπαϊκού εδάφους. Σήμερα η λησαλέα σύγκρουση των οικονομικών συμφερόντων που επέβαλαν μέχρι τώρα αυτή την πολιτική αφήνει γυμνούς τους πολιτικούς ταγούς που την υπηρετούσαν εξοραίζοντας την τραγική πραγματικότητα. Διαπραγματεύσεις χωρίς περιεχόμενο, εκβιαστικά διλήμματα τύπου σχεδίου Ανάν, ανοχή σε δημιουργία τετελεσμένων, παράκαμψη δομικών κανόνων ενταξιακής διαδικασίας ουδέτερες δηλώσεις και συστάσεις για αυτοσυγκράτηση χάραξαν μεταξύ άλλων την πορεία του μπαρμπαρός. Κύριοι συνάδελφοι, είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε το πιο αυστηρό πλαίσιο ώστε να μην επιτρέψουμε την παραμικρή παρερμηνία από κανένα. Οι επιθετικέ ενέργειε τη Τουρκία καταδικάζονται περίφραστα καθώ αποτελούν επίθεση κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των πολιτών τη απειλούν την ενεργειακή ασφάλεια της ένωσης δυναμητίζουν τις προσπάθειες για ουσιαστική λύση στο κυπριακό και επιβάλλουν την επανένταξη της ενταξιακής πορείας της τουρκίας. όποια υποχώρηση από τα Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Σακοράφα και τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό ο συνάδελφος Παπανάκης και στηρίζει τον αγώνα για Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, με μία και μοναδική κυριαρχία, ηθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις, στρατεύματα, ξένους εγγυητές και προστάτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταδικάσει ούτε την τουρκική κατοχή στην Κύπρο, ούτε τις παραβιάσεις της Τουρκίας, ενώ το ΝΑΤΟ προκλητικά συστήνει αυτοσυγκράτηση προς όλες τις πλευρές το κομμουνιστικό κόμμα της ελλάδας απαιτεί την απερίφραστη καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων και είναι αντίθετο με τις προσπάθειες αυτή να υπονομευθεί με τροπολογίες στο ψήφισμα οι οποίες προτάσουν το μοίρασμα των υδρογοναθράκων μεθοδεύοντας μια διχοτομική λύση νομιμοποιώντας τις απαράδεκτες τουρκικές διεκδικήσεις και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της κύπρου και της ελλάδας στη μέγενη των ανταγωνισμών των μονοπωλίων για την ενέργεια συνθλίβεται η δίκαιη επίλυση του κυπριακού. αυτή μπορεί να υπηρετηθεί μόνο σε σύγκρουση με την ευρωπαϊκή ένωση και το νατο με το λαό πρωταγωνιστή για τα δικά του συμφέροντα. ευχαριστώ στον και τώρα ένα η Έχουμε μπροστά μας μια κατάσταση πολύ ενισχυτική. Γιατί, όπως ακούσαμε ήδη από τους συναδέλφους που προηγήθηκαν, αυτή η σωρία απειλών, μονομερών ε, επιθέσεων κατά της Κύπρου, κατά της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, είναι η μεγαλύτερη κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών στο πρόσφατο παρελθόν. Παρά την αναγνώριση της ανταπικής κυριαρχίας από τα κράτη-μέλη που είναι υποχρέωση βάσει του διεθνού δικαίου, υπάρχει ε, ένα σκέλος της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λείπει. Πρέπει λοιπόν να αποστείλουμε στις αρχές της Τουρκίας ένα σαφές μήνυμα και να φανεί αυτό από την τοποθέτηση αυτού του Κοινοβουλίου. Να θυμίσω, όπω ε, εξαιρετικά είπε η συνάδελφος Ελένη Θεοχάρους, ότι έχουμε επανειλημμένως σιωπήσει Έχουμε ανεχτεί στη γειτονιά μας ε, ε, την κατάσταση αυτή που ζει ο Κυπριακός λαός. Πρέπει επιτέλους να ζητήσουμε τη δίκαια λύση με διάλογο και με συνομιλίες. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Γκαρτίνη. Ένα λεπτό, συνάδελφος Μαυρίδης. Πριν μερικέ ώρες γιορτάσαμε την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου. Σήμερα όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα τείχος που επέβαλε ο τουρκικός στρατός και μοιράζει ένα λαό, μία Κύπρο, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους στο ίδιο κράτος. Η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, επιδιώκει με ειρηνικά μέσα να καταργήσει αυτό το τείχος και προσβλέπει στην οικογένεια μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους κανόνες δικαίου. Με βάση λοιπόν αυτό το δίκαιο της θάλασσας μέρος του κοινοτικού ακτιμένου και του διεθνούς δικαίου η κυπριακή δημοκρατία συμφώνησε με όλες τις γειτονικές χώρες αίγυπτο λίβανο και ισραήλ στο διαχωρισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με σκοπό το φυσικό αέριο που προσφέρει προοπτική για ενεργειακή ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ένωση. το ψήφισμα αυτό καταγράφει τα γεγονότα με ξεκάθαρο μήνυμα προς την τουρκία του Ερτογάν να σταματήσει όλες τις παράνομες ενέργειές της εντός της κυπριακής αός όπως επιβάλλουν οι κανόνες δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης. χωρίς σεβασμό σε τέτοιους βασικούς κανόνες δεν μπορεί να λειτουργήσει η ευρωπαϊκή ένωση και επιτέλους η τουρκία ας κάνει το βήμα για σε. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Για ένα λεπτό η συνάδελφος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία γιορτάζει τη νέα στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το νέο σχέδιο δράση το οποίο προτάθηκε. Αλλά αυτό είναι το καινούριο της Τουρκίας και πάλι προκαλεί τη δημοκρατία της Κύπρου και μαζί με αυτήν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει επίδειξη δύναμη. Θέλει τα χρήματα από τα κοιτάσματα. Μπορεί να τα πάρει. Δεν έχει κανεί αντίρρηση, αλλά μόνο αν πάει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όπως ε, ε, η Νότια Κύπρος κάνει υποχωρήσεις. Αυτό δεν ταιριάζει στην Τουρκία, ούτε δεν ταιριάζει όμως και οι άλλες ε, χώρες ε, της περιοχής να μπουν στο παιχνίδι. Το Ισραήλ που και, αυτή είναι, και αυτό είναι αγκάθι στο μάτι της Τουρκίας. Και θέλουμε την ησυχία της να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται το βόρειο τμήμα του νησιού. Και μετά να κατηγορεί την Κύπρο την ε, Δημοκρατία της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν μπορούμε τόσο να αποδεχτούμε. Χρειαζόμαστε καλή σχέση με την Τουρκία, αλλά θα πρέπει να λέμε και τη γνώμη μας στην τελική ανάλυση. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Ζόμερ, και τώρα ένα λεπτό, συνάδελφος Παπαδάκης. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, η κίνηση της Τουρκίας να εκδώσει παράνομη οδηγία ναύτεξ εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλαδή εντός των ευρωπαϊκών συνόρων αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου. υπάρχουν κανόνες δικαίου ή όχι; τελικά επικρατούν τα συμφέροντα στην ευρωπαϊκή ένωση και κλείνουμε τα μάτια; πώς μπορεί η ευρωπαϊκή ένωση να επιτρέπει σε ένα υποψήφιο κράτος μέλος να την εμπέζει και να την κοροϊδεύει με αυτόν τον τρόπο; θέλουμε την τουρκία εντός της ευρωπαϊκής ένωσης όμως δεν μπορεί να γυρνά την πλάτη στι αξίε και στι αρχέ τη Ένωση πρόκειται για μια υποψήφια χώρα που διεκδικεί την έγκριση και τη σύμφωνη γνώμη όλων μας για τη συνέχιση της διαδικασίας. δηλαδή αν δεν τη διεκδικούσε σε ποιες ενέργειες θα είχε προβεί μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει. πώς μπορούμε εμείς να αφήνουμε την τουρκία χωρίς κυρώσεις η οποία με τη δική της ευθύνη απομακρύνεται από τα ευρωπαϊκά θεσμία. Σας ευχαριστώ στον αδελφό Παπαδάκη και τώρα ένα λεπτό στον αδελφό Σπρέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήδη έχουν υποθεί πολλά για το θέμα αυτό και δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία, κράτος ε, μέλος του ΝΑΤΟ, υποψήφια προσένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση πρέπει να δείξει υπευθυνότητα και να αποφύγει μονομερείς ενέργειες οι οποίες είναι απαρέδεκτες. Αυτά που κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα δεχθούμε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κ. Μαυρίδης και να κάνω μια σύγκριση ε, του Κυπριακού με τον ψυχρό πόλεμο, της αντιπαράθεσης Τουρκίας-Κύπρου με τον ψυχρό πόλεμο. Ε, να μην ε, χάνουμε την αίσθηση των αναλογιών δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποια αναλογία μεταξύ των δύο αυτών. Σήμερα είδα με μεγάλη έκπληξη και άκουσα τη συζήτηση για το τείχος ε, του Βερολίνου και την κατάρρευσή του να κάνει τον μεγαλύτερο σε διάρκεια λόγω ένας κομμουνιστής. Έμεινα άναυδος. Και διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφος Καηλή. Αγαπητέ Πρόεδρε, η πτώση του τείχους του Βερολίνου, όπως πολλοί αναφέρανε, δεν επετεύχθη με όπλα, αλλά με γνήσια αλληλεγγύη βασισμένη στο δίκαιο των λαών, τις αρχές της ελευθερίας και την κοινή λογική. Η Λευκοσία όμως, είναι η τελευταία πρωτεύουσα της Ευρώπης με τείχος. αποτέλεσμα στρατιωτική εισβολής και παράνομης κατοχής, κάτι που πρέπει η αλληλεγγύη μας στην Κύπρο να, αναφέρει ρητός να διαφυλάξει την κυριαρχία της και να ασκήσει ελεύθερη τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως κάθε ευρωπαϊκή χώρα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. αλλιώς για ποια ένωση μιλάμε. και εσείς συνάδελφοι στις χώρες σας χωρίς τρομοκρατία και απειλές ασκείτε τα δικαιώματά σας. για ποια ένωση μιλάμε και ποια συμμαχία αν επιτρέπουμε τόση επιθετικότητα εις βάρος μιας χώρας της ευρωπαϊκής ένωσης. Χωρί σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο, η Τουρκία μόνη τη περιθωριοποιείται. Χρειαζόμαστε γεωπολιτική σταθερότητα και να μην συνεχίσουμε τη σιωπή αλλά να έχουμε μια κοινή φωνή ω Ευρωκοινοβούλιο. Και τέλο, είναι αδύνατο να υπάρξει Ευρωπαϊκή Ένωση αν αυτή δεν έχει σύνορα, κοινά σύνορα, το κουράγιο και τη γενναιότητα να τα υπερασπίζεται όταν χρειάζεται από οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη αμφισβήτηση. Σήμερα είναι η Κύπρος, αύριο μπορεί να είναι οι χώρε Βαλτική, μεθαύριο η Φιλανδία. χωρε βαλτικη μεθαυριο η φιλανδια Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό για μια ακόμη φορά μας υπενθυμίζει το υπαρκτό ζήτημα ε, της κατοχής ε, μέρους μιας χώρας μέλους. Ε, δεν ε, πρέπει να δούμε ε, την κίνηση αυτή ε, μόνο ως απειλή για τα οικονομικά συμφέροντα. Είναι και μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Παραβιάζεται και το δίκαιο της θάλασσας, που στόχο έχει ακριβώς την αποτροπή τέτοιων ενεργειών. Τη διαφύλαξη του, της ένομης τάξης, ιδίως από διεκδικήσεις κάποιων χωρών για συγκεκριμένα ύδατα. Η Τουρκία επανειλημμένος έχει δείξει ότι παραγνωρίζει την νομιμότητα της κυπριακής κυβέρνησης. Να λοιπόν μια ακόμη απόπειρα άρνησης και της ίδιας της ύπαρξης ε, της Κύπρου. Εγώ στηρίζω την Κύπρο και καταδικάζω τις ε, συνεχιζόμενες αυτές προκλήσεις της Τουρκίας. Σα ευχαριστώ, συνάδελφε Βαλάσσα. Και τώρα ένα λεπτό ο συνάδελφο Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρόσφατα το τουρκικό σκάφος μπαρμπαρός Οδεία πολεμικών εισέβαλε παράνομα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τη κύπρου με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων. στην τουρκία η κυβέρνηση επιχειρεί την ισλαμοποίηση τη κοινωνία και τον περιορισμό του κοσμικού κράτου στα πλαίσια τη νεοοθωμανική πολιτική τη. η ευρωπαϊκή προοπτική και ο σεβασμό των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή παραμένει η μοναδική πορεία αντίβαρο σε μια τέτοια εξέλιξη και έχει ακόμα σημαντική υποστήριξη στην τουρκική κοινωνία ακριβώς γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση της τουρκίας επιλέγει την όξυνση στην κυπριακή ΑΟΣ. προηγουμένως επέλεξε ατυχώς για αυτήν την πτώση του κομπάνη το ανοιχτό φλερτ με το isis και το πάγωμα των σχέσεων με την αρμενία. σήμερα ζητάμε την αυστηρή καταδίκη των ενεργειών της τουρκικής κυβέρνησης και την άμεση απόσυρση των τουρκικών σκαφών από την ΑΟΣ της κύπρου. στόχος είναι η επανέναρξη των συνομιλιών των δύο κοινοτήτων στην κύπρο για εξέβρεση δίκαιης λύσης του κυπριακού στο πλαίσιο του οηε αυτό είναι ο μόνο τρόπο που εξασφαλίζει τα δικαιώματα των δύο κοινοτήτων στα έσοδα από υδρογονάνθρακα. Σα ευχαριστώ στον Αρφεκύρικο. Ενάμιση λεπτό η κυρία Βόζεμπερκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Χάν, μόλις χθες στη μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας γνωρίζετε ότι εκτενώς συζητήθηκε η παραβίαση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης από την τουρκία σε μια εκτεταμένη συζήτηση. σήμερα η τουρκία παραβίασε επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της ελλάδος πάνω από το νησί μύκονος. σημαίνει αυτό πολύ απλά ότι η τουρκία συνειδητά σε μια στρατηγική επιλεγμένη παραγνωρίζει το διεθνές δίκαιο το κοινωνικό κεκτημένο τη σύμβαση των ηνωμένων εθνών για το δίκαιο της θάλασσας τις αποφάσεις του συμβουλίου ασφαλείας δεν αναγνωρίζει την κυπριακή δημοκρατία δεν σέβεται τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας και διαρωτώ με είπατε στην εισαγωγική σας παρατήρηση ότι περιμένουμε από την τουρκία να δείξει αυτοσυγκράτηση. Άρα άραγε μέχρι πότε; σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Συνάδελφε αποδέχεστε ερώτηση της συναδέλφου Καϊλή. Thank you. Κυρία Βόζεμπερκ, επικαλούμε και την ιδιότητά σας ως δικηγόρου και θα ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η ανοχή του Ευρωκοινοβουλίου και η μη δήλωση, η μη ρητή δήλωση για παράνομη κατοχή στην Κύπρο υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει προηγούμενο που κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στο μέλλον καθώς σήμερα μπορεί να είναι η Κύπρος, αύριο μπορεί να είναι η Βαλτική και μεθαύριο η Φιλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. γνώσεων. Αναμφίβολα είδα την παρατήρησή σας και την εισήγησή σας και συμφωνώ με αυτήν. Το γεγονός και μόνο ότι μια χώρα η οποία διεκδικεί με ενταξιακές συνομιλίες την ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια παράλληλα δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο θα πρέπει αυτό να καθορίσει τη στάση μα να καθορίσει τη στάση μας έτσι ώστε με ψηφίσματα και απλές ανακοινώσεις αποδεικνύεται ότι δεν αποτρέπεται η συμπεριφορά αυτή. Πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί δυνατή και οι αποφάσεις μας να είναι απαγορευτικές πλέον για την ένταξη της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Βόζεμπεργκ. Ένα λεπτό τώρα, ο συνάδελφος Πέγιον. Euh, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τι απογοήτευση είναι αυτή μετά τις ελπίδες που είχαμε το Φεβρουάριο το 2014. Η θέση μας θα πρέπει να είναι σαφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί παρά να καταδικάσει ε, έντονα την παραβίαση των ιδιωτικών δικαιωμάτων και την εισβολή κατά ενός κράτους μέλους. Θα πρέπει να συμφωνήσω απολύτως και με τα λόγια του Επιτρόπου βεβαίως ότι δεν πρέπει να μιλήσουμε για ψυχροπόλεμο ακόμη αλλά να είναι καθαρό το μυαλό μας και να ζητήσουμε ε, απαντήσεις και εξηγήσεις από την Τουρκία. Θα πρέπει και εμεί το ευχόμαστε, η Τουρκία κάποια στιγμή να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεχιστούν οι σχετικέ διαπραγματεύσει. Προκειμένου λοιπόν να δηλητηριάσουμε με δηλώσει την ε, σύγκρουση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, καλό είναι να επιδιώξουμε την ε, ειρήνευση και βάσει του διεθνού δικαίου και για το καλό τη ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και τη Τουρκία. Σα ευχαριστώ, συνάδελφε Και... Ερώτηση, Ερώτηση θέλετε να κάνετε. The question Θέλετε να κάνετε ερώτηση. Επιτρέπετε ερώτηση από τον συνάδελφο. Συνάδελφε Πηγιό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο. Η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται από την δράση του ΝΑΤΟ και η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Εάν όμως καταπατά το διεθνές δίκαιο, μήπως θα έπρεπε να επιβληθούν και ακυρώσεις από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Κύριε Πεγιόν, κοιτάξτε συνάδελφος, κανείς εδώ, και αυτό δείχνει και το ε, πόσο μερικές φορές οι συζητήσεις μας δεν είναι εύστοχες, δεν θα βυσβητήσει το διεθνές δίκαιο. Προφανώς. Όμως, ξέρετε ποια είναι η θέση της Τουρκίας στη γεωγραφική αυτή περιοχή και ξέρετε ποια είναι η στατηγική της θέση. Ξέρετε τι ανησυχίε εγείρονται ούτω ή άλλο σε σχέση και με άλλα ζητήματα, αλλά και με συμπεριφορές της Τουρκίας το τελευταίο καιρό, ιδίως στις ε, συγκρούσεις της ε, Συρίας και του Ιράκ. Θα πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε με σαφήνεια και εντονότατα, αλλά από την άλλη να φροντίσουμε να θερμανθεί ο διάλογος με την Τουρκία. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Πέγιον. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία ΚΑΣΔΙΑ και δυστυχώ δεν μπορώ να επιτρέψω να πάρουν το λόγο πάνω από πέντε συνάδελφοι. Ξεκινάει η συνάδελφος Σπυράκη. Κυρία Σπυράκη. Μικροφόν. Is it working or not? Yes, now. Thank you κύριε πρόεδρε θα ήθελα να θέσω στους συναδέλφους υπόψη τον εξής προβληματισμό το 2004 ήμασταν όλοι σίγουροι ότι η Τουρκία θέλει να είναι υποψήφια χώρα της Ένωσης. Σήμερα, όπως συμπεριφέρεται η τουρκική πολιτική ηγεσία, είμαστε ακόμη σίγουροι το 2014 ότι η Τουρκία θέλει να παραμείνει υποψήφια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα μόνο παράδειγμα θα δώσω από τη μία πλευρά συνεχίζει να αγνοεί δέκα χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις την κυπριακή δημοκρατία. παράλληλα όμως τώρα παραβιάζει εξόφθαλμα την κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη που πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ όλοι ότι είναι η ευρωπαϊκή αποκλειστική οικονομική ζώνη. θέλει λοιπόν η τουρκία να είναι υποψήφια χώρα προς την ευρωπαϊκή ένωση; υπάρχουν τρόποι εκτός από τα ψηφίσματα να στείλουμε ένα σοβαρό ηχηρό μήνυμα προς την τουρκία ότι για να συνεχίσει να διατηρεί το καθεστώ της υποψήφια χώρας θα πρέπει να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. μπορεί αυτό να γίνει ακόμη και με τον περιορισμό της οικονομικής βοήθειας. Α το αντιμετωπίσουμε όλοι εδώ. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Σπυράκη. Και τώρα ο συνάδελφος, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που σήμερα κάνει η Τουρκία, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, προκύπτει από τις δράσεις της στο παρελθόν. Η Τουρκία ε, έχει περάσει με τα στατέματά της σε κατοχή της Κύπρου και έχει φερθεί επιθετικά στις περισσότερες χώρες της περιοχής. Να σας θυμίσω την επιθετικότητα της Τουρκίας προς το Ισραήλ. Να σας θυμίσω τις προκλήσεις της προς τη Βουλγαρία και την Ελλάδα δεν πιστεύω ότι η Τουρκία έχει καμία πρόθεση να συνεχίσει τις καλές προσπάθειες προς την ε, προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σημερινές ενέργειες της Τουρκίας τι δείχνουν. Δείχνουν ότι τέτοιες δράσεις δεν μπορεί να αναλαμβάνει μια χώρα που έχει ευρωπαϊκές προοπτικές. Είναι επιθετική και προκλητική. Καλό λοιπόν όλοι μας να εμείνουμε ε, στο υψηλό στην υψηλότερο επίπεδο να, να, κάνουμε, να απευθύνουμε έκκληση για να πάψει αυτή η επιθετικότητα. Σας ευχαριστώ και τώρα η συνάδελφος Βίκστρομ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Δημοκρατία της Κύπρου έχει το κυριαρχικό δικαίωμα να ασκεί δραστηριότητε στην ε, οικονομική της ζώνη. Αυτό ε, η Τουρκία σε αυτό προκαλεί, που παραβιάζει το διεθνές δικαίωμα. Αυτό πραγματικά είναι ένα τεστ για την Ευρωπαϊκή Ελληνική. Εδώ λοιπόν σήμερα το βράδυ όλοι εδώ σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλοι οι εκλεγμένοι ερετοί θα πρέπει να μιλήσουν με μία φωνή και να σηκωθούν, να ορθώσουν τον αναστημά του, να καταδικάσουν την τουρκική κατοχή τι τουρκικέ δραστηριότητε και να απαιτήσουν η Τουρκία να αποσυρθεί άμεσα. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί απελή για την ασφάλεια όχι μόνο τη δημοκρατία τη Κύπρου, αλλά και για όλη την Ένωση, τη δική μας Ένωση και όλους τους πολίτες μας. Αυτή είναι μια πρακτική που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Βίκστρεμ. Και τώρα ο συνάδελφος Βιέγας. Να ξεκινήσω δηλώνοντας ονόματος της ομάδας μου την ελληνική μου για όσους Κύπριους ζουν, ζουν κάτω από την κατοχή των ε, Ξέρουμε ότι η Τουρκία ε, εισφέβαλε στο βόρειο τμήμα του νησιού, εκτοπίζοντας 10.000 ε, χιλιάδε άτομα. Δεν θα έπρεπε λοιπόν κανείς να ανέχεται τη σημερινή συμπεριφορά της Τουρκίας. Η εισβολή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να την καταδικάσουμε σφοδρά θα πρέπει τα κριτήρια που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση που όταν ε, ακολουθεί τις προσανατολισμούς της Ευρωπαϊκής, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ ε, είναι πάρα πολύ ταχεία στη δράση της, αλλά όχι όταν απειλούνται τα ίδια τα κράτη-μέλη της. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερβεί τον εαυτό της, να καταδικάσει τις ενέργειες της Τουρκίας και να φροντίσει να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με σκοπό την ενοποίηση της νήσου. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Πιέκας. και τώρα τελευταίος στην διαδικασία Καρτιάη ο συνάδελφος Γκρέτσος. Δεν πρόκειται για προκλητικότητα της Τουρκίας. Έχει εισβάλει στο χώρο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και κάνει έρευνες. Πρόκειται λοιπόν για κατάκτηση η ολιγορία όμως που έχουμε επιδείξει ως τώρα απέναντι στις στάσεις της τουρκίας οφείλεται στο γεγονός ότι είναι μέλος του νάτο. εάν δεν ήταν μέλος του νάτο θα ήταν αλλιώτικη η απάντηση η δική μας ενώ της ευρωπαϊκής ένωσης και του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. και αναρωτιέμαι εάν κάτι παρόμοιο έκανε η τουρκία στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία θα ήταν η ίδια η στάση μας. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Καταγγέλλω απερίφραστα την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Επίτροπο, διότι επειδή είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία, γι' αυτό τις θα συγχωρούμε όλα. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Γκλέζη. Τώρα ο Επίτροπος Χάν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στην αποψινή αυτή συζήτηση και σας ευχαριστώ και για τα πολύτιμα σχόλια και επιχειρήματα που προβάλλατε. Πραγματικά είναι πολύ καλό που λάβατε την πρωτοβουλία αυτή για να εκφράσετε την ανησυχία, σα σας για τα πρόσβατα γεγονότα. Θέλουμε και εμείς ε, να εκφράσουμε την ανησυχία μας ε, και να τονίσουμε ε, τις σαφείς υποχρεώσεις που υπέχει η Τουρκία. Είναι ένα μήνυμα το οποίο θα μεταβιβάσουμε στους Τούρκους ζητώντα του τους ε, να προβούν ε, στην εξέβρεση λύσει. Αγαπητοί βουλευτέ σίγουρα πρέπει να βρούμε λύση. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι σε μια εύθραυστη γεωπολιτική κατάσταση και άρα είναι προ όφελο όλων μας ε, να υπάρξει αποκλιμάκωση των εντάσεων και αυτό τάχιστα. Και το συντομότερο δυνατό να υπάρξει πρόοδος και διευθέτηση του Κυπριακού. Νωρίτερα στηρίξαμε την επανέναρξη των ε, διαπραγματεύσεων. Είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι και έτοιμοι να βοηθήσουμε. Τώρα καιρός είναι να δούμε αποτελέσματα και βέβαια πρέπει να στηρίξουμε και τον απεσταλμένο των ΗΕ, τον Έσπεν Μπαρθ Άιντε και τους δύο ηγέτες ε, της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας θα πρέπει να τους συνδράμε στις προσπάθειές τους τώρα που θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια ακόμη φορά και είναι πλέον καιρός να δοθεί μια κατάλληλη απάντηση, η ανδεδειγμένη απάντηση, καθώς επίσης και να δοθεί στήριξη και στις δύο κοινότητες. Ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστώ Επιτροπέ Χάν και τέλος το ψήφισμα Β8 2011-2014 δόθηκε από 7 ε, ομάδες. Αύριο θα γίνει ψηφοφορία. Επόμενο θέμα, η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής ΥΠΑ της Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν. Και θα πάρει το λόγο ο Επίτροπος Χάν, εξ ονόματός της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές. Ε, το Νότιο Σουδάν, η πιο νέα χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι σε πόλεμο, σε πόλεμη κατάσταση επί 11